So, Παρακαλώ τους συναδέλφους αλλά και τους επισκέπτες να καθίσουν. Θέλω να ξεκινήσω την ώρα μου ακόμα και στη τελευταία συνεδρία που θα προεδρεύω, όπως άλλωστε έκανα πάντα. Παρακαλώ τους νέο εκλεγέντες συναδέλφους, τους επανεκλεγέντες συναδέλφους και τους επανερχόμενους. Ε, να καθίσουν. Όπως βέβαια και τους επισκέπτες, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη συνεδρίαση που έχει στόχο τη συγκρότηση της Επιτροπής. Θα εκλέξουμε νέο πρόεδρο και τέσσερις αντιπροέδρους, όπως προβλέπετε από το άρθρο 204 του κανονισμού. Έχουμε πρώτα λοιπόν την εκλογή του Προέδρου και μετά των τεσσάρων αντιπροέδρων. Και τώρα καθήκον μου είναι να σας αναγνώσω τα ονόματα των αντικαθιστωμένων. κυρία Μουσολίνα αντικαθιστά την κυρία Καρνίνη. Ο κύριος Νταχτέν επίσης. Ο κύριος Πίτερλε, τον κύριο Νικολάζετς. Ersetzt durch Sirpa Pitikin, Karl-Heinz Florenz wird ersetzt durch Peter Jahr, Andres Grisip wird ersetzt durch Hoffmann. Das ist die EVP. Αυτό ήταν το ΕΛΚΑ και μετά έχουμε την, τους ελευθέρους Κυρία Ρίς από την κυρία Μάινστερ. ECR. Λίκοφ. Φώστα. Καμάλ. Από τον κύριο Νίκολσον. Και ντόμα. Τον κύριο Τσιμπόνα. Γκουε. Οι εξή αλλαγέ. Ροντρίγκε από την κυρία Κουγιό και η κυρία Αλμαρινά αντικαθιστά επίσης όπως και η κυρία Τέιλερ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σεπτέμβρη. Τα ακούσατε τα ονόματά σας όλοι. Ξέχασα κανέναν, ναι. Έχω κάνει κανένα λάθος. Σιάρς λοιπόν. Dorfman. Dorman. Αντικαθίσατε και δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε για τον αναπληρωματικό. Περνάμε λοιπόν στο κύριο μέρος της διαδικασίας επιλογή, εκλογή Προέδρου. Διαπιστώνω απαρτία του ενός τετάρτου των μελών. 18 ακριβώς συνάδελφοι. Και τώρα πρέπει να δούμε τις προτάσεις για υποψήφιους πρόεδρους. Ο κύριος Λύση έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και θέλω καταρχάς να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους επανεκλεγέντες, νέο εκλεγέντες. Αυτή και μια επιτροπή εδώ, η οποία είχε στην προηγούμενη περίοδο ασχοληθεί με, τις περισσότερες, ε, με τα περισσότερα νομοθετικά ψηφίσματα. Θα συνεχίσουμε πιστεύω την ίδια δουλειά, με την ίδια ένταση. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον μέχρι σήμερα πρόεδρο κύριο Γκρότε και ας μην ανήκει στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έκανε πολύ καλή δουλειά πιστεύω, πολύ σωστή δουλειά. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όμως θέλουμε να υποβάλλουμε υποψηφιότητα για πρόεδρο τον κύριο Τζοβάνι Λαβία, καθηγητή γεωπόνο και πολύ εργατικό βουλευτή σε θέματα και περιβάλλοντος αλλά και ε, γεωργίας ιδιαίτερως αλλά και ε, προϋπολογισμών. Είχε τα θέματα της γεωργίας στον τελευταίο προϋπολογισμό και συμμετέχει μέσω του κόμματός του στην Ιταλία και στην κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να στηρίξει και την Ιταλική Προεδρία και να παρακολουθήσει το έργο της Ιταλικής Προεδρίας και γι' αυτό υποβάλλουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Λαβία. Ευχαριστώ πολύ. Πέτερ δεν βλέπω να έκανε άλλο το λόγο. Ένας λοιπόν ο υποψήφιος μπορούμε να επικυρώσουμε την εκλογή του είτε διαβοής είτε με μυστική ψηφοφορία. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση στην διαβοής εκλογή. Έχει καταθέσει τη δήλωση ε, δημοσιονομικών οικονομικών συμφερόντων ο υποψήφιος και μπορούμε διαβοής να τον επικυρώσουμε και ως εκ τούτου εξελέγει ήδη συγχαρητήρια κύριε Λαβία. Kommen Sie nach oben. Περάστε. Dear colleagues, thank you very much for... Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για την για την εμπιστοσύνη σας. Θέλω να κάνουμε στο δυνατόν καλύτερη δουλειά στην προσεχή περίοδο, θέλω να συνεργαστούμε πολύ καλά όλοι, όλες οι πολιτικές ομάδες για να φέρουμε εις πέρας τη δουλειά που έχουμε για το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν που με εξελέξατε και προχωρούμε με την εκλογή των αντιπροέδρων. Πρώτος αντιπρόεδρος. Παρακαλώ, υπάρχουν υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Κύριε Σάκε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε συγχαρώ καταρχάς για την εκλογή σας. Μη φοβάστε, δεν θα ομιλήσω πολύ. Θέλω να συγχαρώ όλους τους νέους βουλευτές, παλαιούς και εντελώς καινούριους. Νομίζω ότι ε, θα είμαστε απόλυτα δεκτικοί απέναντι σε όλες τις πολιτικές ομάδες και γι' αυτό θα προτείνουμε τον Ούγκρο συνάδελφο Ζάβορ. Δεν Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Τότε με την διαδικασία εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε διαβοής να επικυρώσουμε τον κύριο Ζάβορ στη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. I, I ask Mr. Javor to join us here. Και τον παρακαλώ να έρθει στο Προεδρείο. Now we can go to the second uh, vice chair and... Θέση δευτέρα Πρόεδρου τώρα. Ερωτώ αν υπάρχουν υποψήφοι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρουσιάσω την υποψηφιότητα του κυρίου Βαλεντίνας Ματζουρόνης. Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ματζουρόνη για να παρουσιάσει ο ίδιος την υποψηφιότητά του καλύτερα. Eh, eh, Υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα. Κύριε Χρότε. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες προτείνουν τον κύριο Ζάμπορ που είναι πέντε χρόνια τώρα βουλευτής. Πέντε Έχει εργαστεί στην Επιτροπή αυτή και είναι η πρότασή μας για το δεύτερο αντιπρόεδρο. Okay, Mrs. Hauken, the floor is yours. Yes, I want to take the... Κύριε Hauken. Θα ήθελα να πω ότι εμείς στην πράσινη ομάδα, στην ομάδα των πρασίνων έχουμε μια κάποια δυστημία εδώ να εκφράσουμε ε, υπάρχει μια παλιά πρακτική, εθιμική πρακτική, σύμφωνα με το 199, ε, προσπαθούμε ε, να αντιπροσωπεύονται όλες οι πολιτικές ομάδες ανάλογα με το μέγεθός τους και πρέπει να χρησιμοποιούμε το σύστημα de Hont. Εγώ είναι η τρίτη φορά που εξελέγει βουλευτής και δεν έχω ακούσει κανένα επιχείρημα ε, εναντίον ενός υποψηφίου ο οποίος προτείνεται από την συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, την EFDD. Ε, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούμε η αντιπρόταση δεν είναι σωστή, δεν είναι δίκαιη. Αμαυρώνει τις διαδικασίες ε, τις οποίες ακολουθούσαμε μέχρι τώρα με δικαιοσύνη και ισότητα και αν υπάρχει ε, μια διαμαρτυρία εναντίον ενός υποψηφίου αυτό είναι κάτι άλλο αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι ο υποψήφιος είναι ικανότατος και ο δρόμος ο οποίος φαίνεται να ακολουθείται από αρισμένους είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία στο σύνολο του Κοινοβουλίου. Mr. Θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε η προλαλήσασα, αλλά να το εξηγήσω λίγο. Πράγματι δεν πρέπει να παραβιάζουμε τις συμφωνίες τις οποίες καταλήξαμε, οι οποίες ήταν μακρόχρονες και περίπλοκες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε η μία ομάδα την άλλη, γιατί αν πραγματικά θέλουμε να σπάσουμε το σύστημα, τότε ε, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Όμως θα ήθελα εδώ να διευκρινίσω κάτι, επί τη βάση αυτών που είπε η κυρία Άουγκεν. Ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ οι πράσινοι επιτέθησαν για να μην δώσουν την δυνατότητα να πάρει η θέση αντιπροέδρου το μέλος ε, της ECR. Οπότε η στάση σας είναι υποκριτική. Σας στηρίζω αλλά υποστηρίζω ότι η στάση σας είναι υποκριτική με βάση αυτά τα οποία είπα στην αρχή, αλλά βέβαια η υποκρισία δυστυχώς σύνορα δεν έχει. Ε, ε, ε, λάθος πινακίδα δεν είμαι ο κύριος Σπότς, κύριε Λαβία. Λάινεν. τρέφω μεγάλη εκτίμηση προς την κυρία Άουκεν. Έχουμε εργαστεί πολύ καλά τελευταία πενταετία. Μάργκρετ, είπε ότι σε τρει ε, θητείε εδώ στο Κοινοβούλιο, εγώ τέσσερι πάλι και έχω δει αρκετέ φορέ να μην εκλέγεται κάποιο για διάφορου λόγου που έχουν να κάνουν και με την ομάδα του. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο αυτό. Έχει συμβεί αρκετέ φορέ. Και έχουμε ασφαλώ σοβαρότατου λόγου για του οποίου προτείνεται μια άλλη υποψηφιότητα στην ε, θέση αυτή. Κύριο Λίσσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πρέπει να κάνουμε μια πολύ προσεκτική διάκριση μεταξύ των προσωπικών και των πολιτικών λόγων. Εδώ η Επιτροπή αυτή είναι ένα πολιτικό όργανο, δεν έχει να κάνει λοιπόν η επιλογή με την προσωπική ακαιρεότητα του υποψηφίου της ομάδας FDDD, αλλά με την ομάδα την ίδια. Το σύστημα DONT δεν είναι θεόπεμπτος κανόνας, βοηθάει για την κατανομή των θέσεων, αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα κριτήρια για την απόφαση του ποιο θα είναι πρόεδρο και αντιπρόεδρο σε μια επιτροπή, κάτι το οποίο έχει συμβεί και με σύμπραξη των Πρασίνων κατά την εκλογή σε διάφορε θέσει του Κοινοβουλίου. Την προηγούμενη εβδομάδα. Από κοινού, αν δεν απατώμε και με ψήφου των Πρασίνων δεν δώσαμε θέση αντιπροέδρου σε εκπρόσωπο του FDD αλλά σε έναν δεύτερο φιλελεύθερο υποψήφιο πράγμα το οποίο επίσης παραβίαζε το σύστημα DONT. Άρα το επιχείρημά σας δεν ε, ευσταθεί. Η δε ομάδα FDD θα πρέπει να αποφασίσει είτε θα στρέφει τα νότα της την ώρα που ανακρούεται το Ευρωπαϊκό Σύμνος, πράγμα το οποίο έχει πολιτικές συνέπειες, αν του ποιος είναι υποψηφιός της. Εξού και εγώ ε, υποστηρίζω την υποψηφιότητα της κυρία Ζάμπου με μεγάλη εμπειρία όλα αυτά χρόνια, πολύ επιμελή δουλειά στην Επιτροπή μας και ως εκ τούτου για μένα μια εξαίρετη υποψήφια. Κύριε Άουκεν, θα ήθελα να πω ότι όταν καταψηφίσαμε προτινόμενο υποψήφιο, το πράξαμε λόγω της ε, απουσίας κάποιων ικανοτήτων ή δεξιοτήτων στο πρόσωπό του. Και ως εκ τούτου η επιχειρηματολογία μας στηρίζεται στο πρόσωπο και όχι στην ομάδα. Το να αξιοποιείται λοιπόν τέτοιο επιχείρημα κατά μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός δεν το καταλαβαίνω. Αν είχατε κάποια επιχειρήματα κατά κάποιου υποψηφίου, αν θεωρούσατε ότι ένα συγκεκριμένο υποψήφιο δεν θα μπορεί να ηγηθεί των εργασιών τη Επιτροπή κατά επαρκή τρόπο, θα το δεχόμουν. Αλλά ε, μια ομάδα ή ένα πολιτικό κόμμα να το αποκλείεται λέγοντας ότι δεν μα αρέσει και διαφωνούμε μαζί του, το βρίσκω και ανέντιμο και αθέμητο σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Ποιος άλλος ακόμη θέλει το λόγο. Μίστερ Μαζουρόνης. Ο κύριος Ματσουρόνης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιαστώ. Λέγομαι Βαλεντίνος Ματσουρόνης. Ήμουν υπουργό ε, Περιβάλλοντος στη Λιθουανία. και μάλιστα είχα προεδρεύσει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εδώ και έξι μήνες τελείωσε η προεδρία μας. Η εμπειρία την οποία συνέλεξα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της χώρας μου στο Συμβούλιο, η συνεργασία με τους επιτρόπους, με τους συναδέλφους στο Συμβούλιο, και φυσικά η εμπειρία της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου ήταν όλα πάρα πολύ χρήσιμα και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι η εμπειρία αυτή θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε όλους. Αλλά όλα φυσικά θα εξαρτηθούν από τη δική σας ψήφο, από τη δική σας επιλογή και απόφαση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων Υπάρχουν ισορροπίες στο εσωτερικό των ίδιων των πολιτικών ομάδων, ανεξαρτήτως όμως της συγκεκριμένης δυνατότητας επιλογής, αν με υπερψηφίσετε, ε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας και θα μπορέσουμε να επιλέξουμε τις καλύτερες λύσεις για τους πληθυσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να πάρετε τη σωστή απόφαση. Much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάρμπου για να κάνει και τη δική της παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους λοιπόν και αυτού που με υποστηρίζουν και αυτού που δεν με υποστηρίζουν. Η δεύτερη μου θητεία στην Επιτροπή αυτή. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο τη Επιτροπή αλλά και με τους τη της ε, Επιτροπής, του βουλευτέ. Η εμπειρία που έχω συλλέξει από την Επιτροπή περιβάλλοντο, αλλά και πέραν αυτή η εμπειρία που έχω συλλέξει στην ίδια τη Ρουμανία κατά την ε, ενασχόλησή μου με τις οργανώσει οργανώσεις στον χώρο του περιβάλλοντος ε, με οδηγούν σε στη διαπίστωση ότι καθώς είμαστε εδώ ως πολιτικοί που μας έχουν αποστείλει οι ψηφοφόροι μας, θα πρέπει και να τους εκπροσωπούμε. Δεν πρέπει να λησπολνούμε δηλαδή ότι εκπροσωπούμε είτε μέσα στην Επιτροπή είτε στην Ολομέλεια τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα λοιπόν της οποίας είμαι μέλος και της οποίας ε, και την οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντική Ναι. Νομίζω ότι μου δίνει το δικαίωμα να είμαι υποψήφια. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σα. Uh, uh, λοιπόν, θα πρέπει να ψηφίσουμε. Όταν έχουμε δύο υποψηφίους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υποχρεωτικά την ηλεκτρονική κάρτα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Αν θέλετε να ψηφίσετε τον κύριο Ματσουρόνης, θα πρέπει να πατήσετε το πράσινο κουμπί. Αν θέλετε να ψηφίσετε την κυρία Σάρμπου θα πρέπει να πατήσετε το κόκκινο κουμπί. Πράσινο για Ματσουρόνης και κόκκινο για την κυρία Σάρμπου. Λοιπόν, έχετε όλοι τις κάρτες σας. Μήπως έχει ξεχάσει κάποιος. Κοιτάξτε, έχω ξεχάσει την κάρτα μου, λέει ένας ε, Okay. the problem with uh, a λοιπόν, λύθηκε το πρόβλημα. Θα υπάρξει κάποιος αναπληρωτής φορέντσα που θα πάρει μέρος στην ψηφοφορία. Είπαμε ματσουρώνεις πράσινο κουμπί, Σάρμπου κόκκινο κουμπί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Oh. We have one EPP. Ε, από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο υπάρχει μία επιπλέον ψήφο. No, no, only one. Μία ψήφο επιπλέον. Okay. We close the vote. Πέρα τη ψηφοφορία. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. We have. Uh... Oh, ah, yes, Okay. Λοιπόν, δεύτερος αντιπρόεδρος η κυρία Σάρμπου. Ζητώ από την κυρία Σάρμπου να ανέβει στο Προεδρείο. And now we are going to vote for the... Τώρα ε, θα ψηφίσουμε για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Okay, Mr. Gott, the floor is yours. Ich schlage Pavel Potsch. Προτείνω τον Παύλ Πότς. Ο Παύλ Πότς δεν είναι ο Γιολάινεν. Είναι μέλος της Επιτροπής μας εδώ και πέντε χρόνια. έχει παρακολουθήσει σοβαρές ε, διαδικασίες νομοθετικές, έχει μεγάλη εμπειρία και είναι η δική μας πρόταση για τρίτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής. We have other Υπάρχει εδώ τώρα άλλη υποψηφιότητα. Όχι από ό,τι φαίνεται. Έχω εδώ την δήλωση του κυρίου Πότσου αποδέχεται την υποψηφιότητά του οπότε μπορούμε ε, να υπεψηφίσουμε διαβοής, να ψηφίσουμε διαβοής, συγγνώμη. Ε, εξ ονόματος της EFDD θέλω να προτείνω τον κύριο Φρόντ Uh, θα μιλήσω Ιταλικά γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω εύκολα. Το αίτημα να, πάρει το λόγο ο συνάδελφος έγινε ταυτόχρονα με, την, με το αίτημα το δικό μου για την ψηφοφορία διαβοής. Αν επιμένει για την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Φυσικά επιμένω οπότε θα πρέπει να ψηφίσουμε για μια ακόμη φορά με την ηλεκτρονική κάρτα. Με το ίδιο σύστημα, δηλαδή αν θέλετε να υπεψηφίσετε τον κύριο Φρόντε θα πατήσετε το πράσινο κουμπί. Αν θέλετε τον κύριο Πότς θα πατήσετε το κόκκινο. Πράσινο Φρόντε, κόκκινο Πότς.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 Τέλος της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι το εξής, 42 για τον κύριο Πότς και 19 για τον κύριο Φρόντε. Συγχαρητήρια στον κύριο Πότς λοιπόν, ο οποίος δεν είναι παρόν. Και περνάμε τώρα στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Κύριε Χρόντε. Schlage Gilles Προτείνω το Σιλπανιού. Συνάδελφο με μεγάλη εμπειρία εδώ στην Επιτροπή. Έχει εργαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια και τον προτείνουμε ως τέταρτο αντιπρόεδρο. Ζητούμε λοιπόν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων. Mr. Νίκολσον. Μιας και τα πράγματα πήγανε όπως πήγανε, εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα σε αυτό το βαθμό. Προτείνω λοιπόν την κυρία Τζούντιθ Γκάρλιν, που ήταν τα τελευταία πέντε χρόνια μέλος της Επιτροπής μας. Okay. See, uh... Μάλιστα. Και εγώ είμαι νέος και δεν έχω δει ξανά μια τέτοια κατάσταση και γι' αυτό θέλω να παρουσιάσω μια νέα υποψήφια του EFDD, την κυρία Εύη. Avendo e trovandoci Τώρα λοιπόν έχουμε τρεις υποψηφιότητες. Ε, σε αυτή την περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι η ψηφοφορία να γίνει πάλι με την κάρτα. Και γι' αυτό έχουμε τρεις υποψηφίους όπως είπα. Τον κύριο Παρνιό, την κυρία Γκέρλινγκ και την κυρία Λέβη και γι' αυτό διακόπτουμε για λίγα λεπτά έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι κάρτες. η διανομή των ψηφοδελτίων θα, σας αρχίσουμε, θα αρχίσουμε να σας φωνάζουμε. Να πω ότι ορισμένοι συνάδελφοι επιγόντως πρέπει να πάνε και σε άλλες επιτροπές και γι' αυτό παρακαλώ να τους φωνάξετε κατά προτεραιότητα γιατί πρέπει να πάνε να ψηφίσουν και αλλού.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 Sciulza. Questa? Oh? Onecka. Dov'è Onecka? Onecka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign.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

Οκ. Okay. Ωραία. Θα ανακοινώσουμε τα Number of voters 63. 63 εψήφισαν. Τρία λευκά. 60 έγκυρα. Απαιτούμενη πλειοψηφία 31. Παρνιό 37 Αρνιό. Γκίρλινγκ 12 και Χέβι 11. Απομένως ζητώ από τον κύριο Παρνιό να έρθει να καθίσει εδώ στα Προεδρία. Now we can go to the third point. Τώρα το τρίτο σημείο. ανακοινώσει του Πρόεδρου. Πρώτον, ακρόαση της υποψηφίας Επιτρόπου Φερότσι. Μετά την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της 3ης Ιουλίου για τη διαδικασία αυτή για την αντικατάσταση των Επιτρόπων, Η ακρόαση της υποψηφίας Νέλη θα οργανωθεί από την Επιτροπή Ήτρε την Δευτέρα 14 Ιουλίου στις 12.30. Επειδή είναι πολύ σύντομος ο χρόνος που μένει μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Κομισιόν και επειδή δεν θέλουμε να υπάρξει επικάλυψη με τους επόμενους επιτρόπους, η διάσκεψη των Προεδρών αποφάσισε να εφαρμόσει μια ελαφρύτερη διαδικασία από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για τις ακροάσεις της δεύτερης επιτροπής Μπαρόσο το 9. Επομένως, επειδή είναι πολύ λιγότερος ο χρόνος που έχουμε για κάθε ακρόαση, μόνο τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση της Ήτρε, θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα στον υποψήφιο επίτροπο. Παρ' όλα αυτά θα είναι δημόσια η συνεδρίαση και τα μέλη της Επιτροπής Περίφ καλούνται να παραστούν. Η συνάντηση αυτή τη Ήτρε, σα επανθυμίζω, είναι 14 Ιουλίου στις 2.30, Δευτέρα. Δεύτερη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμά μας. Λόγω του άχθους της εργασίας, νομοθετικής εργασίας στην αρχή της θητείας, η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει 21 και 22 Ιουλίου και θα τελειώσει την 5η στις 12.30, 24 Ιουλίου. Όχι το απόγευμα όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Το χρονοδιάγραμμά μας μέχρι το τέλος του χρόνου θα εγκριθεί από τους κοσμήτωρες στην πρώτη του συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου το απόγευμα σας υπενθυμίζω θα γίνει η παρουσίαση της Ιταλικής Προεδρίας των Προτεραιοτήτων της από τους Υπουργούς Γκαλέτη και Λορεντζίν και θα αρχίσει στις 9 εδώ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 23 Ιουλίου. Αυτά για σήμερα και σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας.